Okay, Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι. Έχουμε έναν πολύ νεαρό Ευρωπαίο πολίτη παρόντα στην αίθουσα. Είναι ο πιο όμορφος Ευρωπαίος πολίτης που έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Οι σοσιαλιστές έχουν μία ψήφο παραπάνω χάρη σε αυτό το παιδάκι. Το αξίζουν νομίζω. Ας είμαστε λοιπόν πολύ καλοί τώρα που έχουμε την παρουσία ενό τόσο νεαρού Ευρωπαίου πολίτη. Λοιπόν, ας περάσουμε στην συνάντηση των ε, συντονιστών, να σας ενημερώσω. Πρώτα απ' όλα είχαμε τα θέματα 9 και 10 Νοεμβρίου εγκρίθηκαν και οι συντονιστές συμφώνησαν για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 που δόθηκε στους σοσιαλιστές. Και για το Μαρακές η υπεύθυνη είναι η Γιούρη και εμείς συμφωνήσαμε για γνωμοδότηση επί του κανονισμού που ανατέθηκε στο ΕΛΚ. Α, όχι. Στους πράσινους διορθώνει η Πρόεδρος. Και η οδηγία ανατέθηκε στο ΕΛΚ. Οι συστάσεις συγκρίθηκαν, όπως τις πρότεινα εγώ, με κάποιες προσθήκες και κάποιες διορθώσεις. Τώρα για τα διάφορα έτοιμα γραπτά θα σας ενημερώσουμε γιατί υπήρξαν τόσα πολλά θέματα που θα έπρεπε να τα δείτε όλα. Τώρα επίση. Ενημέρωσα τους δωνιστές ε, για δύο θέματα προφορικά. Για τη συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την ακρόαση που είχαμε τον Ιούνιο. Και ενημέρωσα και για τη συνάντηση με τους ε, επιτρόπους, στο Σώμα των Επιτρόπων που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο. Τώρα για τις ακροάσεις και τις ερευνητικές ε, αποστολές όσον αφορά το πρώτο εξάμενο του 2017, αποφασίσαμε να έχουμε μία μίνι ακρόαση με την ΛΥΜΠΕ για τους απάτριδες και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και σε βάρος των ανηλίκων. Θέματα τα οποία αναφέρονται σε αναφορές που μας φτάνουν μετά από διάφορα γεγονότα και διάφορων μορφών διακρίσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συμφωνήσαμε αυτό, όπως επίσης και την ε, εμπιστοσύνη των πολιτών, πώς θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και αυτό συμφωνήθηκε από τους συντονιστέ. Οπότε προσβλέπουμε στις ακροάσεις αυτές στις αρχές του 2017. Αποφασίσαμε Επίση, να έχουμε και μια επίσκεψη στην Ισπανία ερευνητική για τα χαμένα παιδιά. Και στην Σουηδία για το θέμα του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης που έχουμε στην Σουηδία και που μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να το αποκτήσει κανείς, ιδιαίτερα όταν έχουμε διασυνοριακά ζητήματα και ακόμα πιο δύσκολο για τα παιδιά. Οπότε πρέπει να μάθουμε περισσότερα. Για την υδρορογμάτωση τώρα. Έχουμε τέτοιες αναφορές που έχουν ήδη συζητηθεί τον Ιούλιο και σε συνέχεια αυτών οι συντονιστές αποφάσισαν να συντάξουν γνωμοδότηση εφόσον υπάρξει έκθεση πρωτοβουλίας είτε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος είτε από την Ήτρε. Για το πόρταλ της Επιτροπής μας Αναφορών αποφασίσαμε Απλώς ενημέρωσα και είπα ότι όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να απευθυνθεί στη γραμματεία. Αυτά περί συντονιστών. Και συνεχίζουμε με τη σημερινή μας ημερήσια διάταξη και πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε για την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο 2015. Ελπίζω να έχετε βάλει όλοι στο μηχάνημα τις κάρτες σας, σωστά. Οπότε ψηφίζουμε. Συμβιβαστική τροπολογία α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Α, καταπίπτει. Έχετε δίκιο. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της προφορίας. Διακόπτη. Δεν ψηφίσατε. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί. Η κάρτα. Ωραία, τότε θα πρέπει να μας λέτε. Με το χέρι σας, έτσι, διανατάσσεως της χειρός. Έτσι κι αλλιώς εγκρίθηκε η τροπολογία. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία Γ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σαράντα πέντε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σαράντα έξι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία δέλτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, όχι, 68 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τώρα συμβαστική τροπολογία F, F, σιγματάφ, F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, όχι, 77 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79. Θέλετε να ελέγξουμε για την 78. Ωραία, θα παληθεύσουμε. 78 τροπολογία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. 79 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται. Εγώ το είπα λάθος, λέει πρόεδρος. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε, αλλά να ελέγξουμε, να επαληθεύσουμε για να είμαστε σίγουροι. 81. Ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε βέβαια. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, θα επαληθεύσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική I για υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να παληθεύσουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 101. Ψηφίστε. Πέρα τη φοφορίες, εγκρίθηκε. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 2 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αριθμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ,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 Συμβαστική τροπολογία J υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία τώρα, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας της ε, ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην ψηφοφορία. Μην ξεχάσετε τις κάρτες σας ε, στο μηχάνημα. Νομίζω ότι αρκετοί δεν θα παραμείνουν στην αίθουσα, άρα ας αποχωρήσουν διακριτικά και οι υπόλοιποι καθίστε. So, the next... Το επόμενο θέμα είναι η διερευνητική επίσκεψη στη Σλοβακία 19 με 23 Σεπτεμβρίου. 19 με 22 Σεπτεμβρίου φέτος. Λίγες εβδομάδες πριν. Πρόκειται για μια προφορική έκθεση και αργότερα θα καταρτήσουμε μια έκθεση. Θα ήθελα να σας πω ορισμένα λόγια. Δηλαδή φτάσαμε στη Μπρατισλάβα, είχε γίνει μία αναφορά που είχαμε λάβει το 12 με μία συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάσαμε αυτή την ε, έκθεση σε σχέση με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων σε ε, διάφορα ε, κέντρα κατοικίες για άτομα με αναπηρία στη Σλοβακία. Μπορώ να πω ότι υπήρξε μεγάλη συνεργασία από τους εμπλεκόμενους φορείς, της ΜΚΟ, τις κυβερνητικές αρχές και τους ανθρώπους, το προσωπικό που διαχειρίζεται την κατάσταση κάθε μέρα. Επισκεφτήκαμε τρία κέντρα, ένα κέντρο ε, ημερήσιας ε, φροντίδας, ένα άλλο κέντρο για αμαία όπου είδαμε πώς μπορεί να... Ε, πώς μπορεί, μάλλον πώς είναι η καθημερινή ζωή σε αυτά τα κέντρα. Ε, εδώ έχουμε και 130, σε αυτό το κτίριο είχαμε 130 ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτό το κέντρο σε, για όλη τους τη ζωή. Οι ΜΚΟ μας είπαν ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί με αναπηρίες να μην ε, πάσχουν από ιδρυματισμό. Φυσικά θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη πρόοδος η πορεία είναι πολύ αργή, γι' αυτό θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα από τους άλλους, να είναι αυτόνομοι και αυτοεξυπηρετούμενοι. Τον Ιούλιο ανέκυψε νέα νομοθεσία έτσι ώστε τα ΑΜΕΑ να έχουν ε, και δικαιώματα τα οποία να καλύπτονται νομικά. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Και αντιβαίνει με το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των ΑΜΕΑ. Επίσης, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να διασφαλιστεί. και για να έχουν πρόσβαση και στην αγορά και στη, ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας και να απομακρυνθούν από αυτό το καθαρά ιδρυματικό πλαίσιο στο οποίο ε, λειτουργούν. Δυστυχώς μέχρι τώρα μόνο το 10% των 861 Ιδρυμάτων στη Σλοβακία έχουν ενταχθεί στην κοινωνική ζωή. Ως προς ε, την συμμετοχή αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση από τις κρατικές αρχές για να μπορούν να ε, είναι αυτόνομοι και αυτοεξυπηρετούμενοι Δηλαδή θα πρέπει να ισχύει το nothing about us without us. Θα μπορούσα να μακρηγορήσω βεβαίως, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει ευθύνη με βάση ε, λοιπόν τα στοιχεία των ΜΚΟ μπορεί να επέλθει πραγματική ε, αλλαγή για να γίνει σωστή χρήση των διαρθρωτικών όρο. Και για να απομακρυνθούν από αυτή την κατάσταση ιδρυματισμού, να επανενταχθούν στην κοινωνία οι άνθρωποι αυτοί. Να γίνει η αποϊδρυματοποίησή τους. Η Σλοβακική κυβέρνηση θα μας ε, πληροφορεί γραπτό σε τακτά χρονικά διαστήματα για όλες τις εξελίξεις από ιδρυματοποίησης, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να ενταχθούν στην ενεργό ζωή. Αυτή τη στιγμή η έκθεση θα συζητηθεί στην Επιτροπή τον Νοέμβριο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήρθαν μαζί μας στη Σλοβακία και να ευχαριστήσω και την συνάδελφό μας, τη Ρίτα από τη Γραμματεία, η οποία μας βοήθησε ιδιαίτερα και εκεί και στην κατάρτιση της έκθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Παλ που μας βοήθησε για να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς που έπρεπε και να έχουμε και μία να δούμε και την Πρατισλάβα που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή πόλη. Τώρα, λοιπόν, ε, σας δίνετε ευκαιρία να επισκεφτείτε την πόλη υπό Σλοβακική Προεδρία. Τώρα, θα στραφούμε στην αναφορά στο σημείο 17.06.94 του 15 της Ευστρατείας Καμπούρη με 108 υπογραφές σχετικά με τις παραβιάσεις δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων κατά την ανάθεση της Σύμβασης Αξιοποίησης Μεγάλης Έκτασης στην Αττική, το πρώην αεροδρόμιο ελληνικό. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Δίνω το λόγο στην αναφέρουσα. Σας καλωσορίζουμε και έχετε το λόγο. Ναι. Ε, καλησπέρα σας. Ε, είμαστε δύο εδώ αναφέροντες. Σας είχα ενημερώσει, μου είχατε πει να σας ενημερώσω μέχρι τις 28 Σεπτέμβρη, οπότε και ενημέρωσα ότι θα είμαστε δύο. Okay. Θα σας δώσω πέντε λεπτά για δύο. Δυόμιση και δυόμιση. Ωραία. Ξεκινάω εγώ. Εντάξει. Α, όχι, ξεκινάει ο κύριος Πρασάς, ο οποίος είναι εκεί. Ναι, εντάξει. Θα, θα αρχίσετε εσείς. Ο λόγος είναι για σας. Καλησπέρα. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Η αναφορά μας ε, αφορά την εκποίηση δημόσιας ε, παράκτειας έκτασης 620,6 εκταρίων παραλίας 3,5 χιλιόμετρων που βρίσκεται στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Αυτή η εκποίηση είναι ένα σκάνδαλο και πολιτικό και οικονομικό και περιβαντολογικό. Το 2010 με την είσοδο της χώρας μας σε καθιστός οικονομικής επιτήρησης, το ελληνικό εντάχθηκε στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης με όρους επαχθής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σημασία του για μια περιβαντολογική ανάταση του λεκανοπεδίου. Να, θεωρεί, να καταλάβουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Στην Αθήνα υπάρχουν 2,5 τετραγωνικά πρασίνου ανακάτοικο αντί για 12 που είναι τα διεθνή standards. Το τίμημα της πώληση είναι 915 εκατομμύρια σε βάθος δεκαετίας, ενώ άμεσα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 574 εκατομμύρια. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος εκτίμησε ότι το τίμημα αυτό θα έπρεπε να ήταν στα 3 δις και δύο εμπειρογνώμονες που όρισε ο Ισαγγελίας διαφθοράς σε 1,5 και 2,3 δις. Θα με συγχωρέσετε γιατί πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κάνω ε, μία αναφορά και θα ήθελα πραγματικά το να μπορέσετε να έρθετε στην Αθήνα για να, να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής που θα συντελεστεί εάν και εφόσον προχωρήσει το συγκεκριμένο project. Η παραβίαση του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, καθώς και η παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης του ανταγωνισμού, οι οποίες διέπουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν συντελεστεί στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, οι τροποποιήσεις των όρων της σύμβασης που θα περιγράψουν παρακάτω γύρουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων υπέρ του επιλεγέντος αγοραστή, επειδή παρέχει πλεονέκτημα στον τελευταίο, με την, ευρωπαϊκή, ε, με την ευνοϊκή μεταχείρισή του, ικανή να νοθεύσει τον ανταγωνισμό. Ακόμα γύρουν θέματα παραβίαση των αναρχών διαφάνεια τη ίση μεταχείριση του ανταγωνισμού, καθώ καμία από τι παρακάτω προβλέψει δεν περιλαμβάνεται στην αρχική προκήρυξη και τροποποιήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν ήταν πλέον δυνατή η υποβολή προσφορά από άλλου ενδιαφερομένου. Η παραχώρηση στον, στον αγοραστή του δικαιώματο επιφάνεια για 99 έτη και το 30% εξαδιαιρέτου πλήρου κυριότητα των εκτάσεων. Η παραχώρηση στον αγοραστή του 100% των μετοχών της εταιρείας, της εταιρείας ελληνικό ΑΕ κατ' υπέρβαση της προκήρυξης, η οποία προβλέπει την παραχώρηση 70% των μετοχών, ενώ το 30% παραμένει το δημόσιο. Οι φοροαπαλλαγές βάσει της υπαγωγής της επένδυσης για το έργο στη διατάξεις του νόμου 2687 του 1953 παρακαλώ ο οποίος μεταξύ των άλλων τις προβλέπει βέβαια. Θεσμοθέτηση νομοθετικής πράξης με την οποία θα συστήνεται φορέας επιφορτισμένος με τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων. Περιέχει φωτογραφική διάταξη με την οποία παρέχεται στον αγοραστή άδεια καζίνο μέσω ενός δίθεν δημόσιου διαγωνισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 8 προβλέπεται αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του δημοσίου που θα στεγαστούν. Το αντίτιμο που θα πληρώσει το δημόσιο για τις 300.000 τετραγωνικά μέτρα για χρήση κοινή ωφέλεια θα είναι τεράστιο. Παράλογα και χαρακτηριστικά δικαιώματα στον, του αγοραστή για αποζημίωση σε περίπτωση που υπάρχει. Ανακάλυψη αρχαιοτήτων στο υπέδαφο καθώ και στον θαλάσσιο χώρο. Σημειωτέων στο συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται τρει αρχαίοι δήμοι από ό,τι βλέπω ο χρόνος έχει περάσει. Θα με συγχωρέσετε που δεν μπορώ να αναπτύξω παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και, και τώρα ήρθε η ώρα για, για κυρία Καμπούρη. Ναι. Ο λόγος είναι για σας. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, εξαιτία του, του χρέους η χώρα μας υποχρεώνεται στη συστηματική παραβίαση του νοσιακού δικαίου. Πρόσφατα, προαπαιτούμενο των δανειστών ήταν και η ολοκλήρωση της πώληση του ελληνικού η οποία βρήθη παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου και συγκεκριμένα. Παραβιάζεται η Οδηγία 2001 και η Διεθνή Συνθήκη του Άρχους και αναφέρουμε συγκεκριμένα πώς παραβιάζεται. Επιλέγει ένας νόμος, η οδός της παράκαμψης, δηλαδή της πάγιας χωροταξικής και πολυδομικής διαδικασίας στην πατρίδα μου και το σχέδιο αξιοποίηση του ελληνικού περιελήφθη σε ειδικό νόμο, ενώ έπρεπε να είναι διοικητική διάταξη. Αυτό έγινε γιατί δεν θα μπορούσε να βγει διοικητική διάταξη, διότι θα ήταν παράνομη, διότι δεν το προέβλεπε το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, που είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός. Όμω, το γεγονό ότι το σχέδιο ανάπτυξη του ελληνικού δεν αποτελεί διοικητική πράξη, προβλεπόμενη από νόμο, όπω λέει η Κομισιόν, αλλά έχει συσπιστεί από ειδικό νόμο, δεν απαλλάσσει το ελληνικό δημόσιο από την υποχρέωση συμμόρφωση με την οδηγία διότι υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε 287 κάθετος 98 που έχει αποφανθεί επ' αυτού. Επιπλέον, οι ρυθμίσει του νόμου αυτού του 4062 είναι συγκεκριμένε και δικέ. Καθορίζουν χρήσει γη, όρου και περιορισμού δόμηση, οι οποίε δημιουργούν αυτή καθ' αυτή και το πρώτον σοβαρού κινδύνου για το φυσικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, τι ακτέ και τη βιοπικιλότητα. Συνεπώ, η διαδικασία τη στρατηγική περιβαλλοντολογική εκτίμηση που προβλέπει η οδηγία έπρεπε να προηγηθεί τη ψήφιση του νόμου τότε που το σχέδιο ήταν υπό ανάπτυξη, δηλαδή σε προθύστερο χρόνο, επειδή ήταν ο κατάλληλο χρόνο για να εξεταστούν οι εναλλακτικέ λύσει συμπεριλαμβανομένη και τη μηδενική και να εκτιμηθούν οι επιπτώσει του και η ενημέρωση και διαβούλευση με το κοινό. Ε, παραβιάζεται επίση η Οδηγία 92 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώ οι προβλεπόμενε επεμβάσει στην ακτογραμμή, έχει μια ακτογραμμή 3,5 χιλιόμετρων αυτή η περιοχή, η αλλαγή χρήση γη θα καταστρέψουν σημαντικού βιότοπου με λιβάδια Ποσειδονία, τα οποία ανήκουν στα είδη προτεραιότητα για τη διατήρηση των οποίων η κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη. Έχει και υφάλου με κοριαλογενεί σχηματισμού. Σα είχα στείλει ένα βίντεο και θα σας το καταθέσω κιόλας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών αναφέρει σε έκθεσή του ότι τα στοιχεία της βιοπικιλότητας του θαλασσίου οικοσυστήματος στο ελληνικό αρκούσαν για να ενταχθεί η περιοχή αυτή στο δίκτυο Natura και φυσικά μόνο έχουν ενταχθεί 6,5% στο δίκτυο Natura σήμερα στο, στο θαλάσσιο χώρο. Παρ' όλα αυτά, η έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, αναφέρει ότι η περιοχή αυτή είναι biodiversity hot spot Οπότε πρέπει να προστατευτεί. Επίσης αντίκειται ο νόμος αυτά που, θα, που προβλέπει και στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία 2060, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη πρέπει να επιτύχουν καλή οικολογική ποιότητα σε όλα τα υδάτινα σώματα έως το 2002. Το ΕΛΚΕΘΕ λοιπόν πάλι στην έκθεσή του δηλώνει ότι οι επεμβάσεις στο ελληνικό θα υποβαθμίσουν την ε- οικολογική ποιότητα του εσωτερικού σαρονικού με αποτέλεσμα η χώρα να μην εκπληρώσει το στόχο. Τρίτη παραβίαση είναι η παραβίαση της συνθήκης Φλωρεντίας για το τοπίο. Εκεί θα δομηθούν 3 με 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, 16 όραφα ακτήρια, 7 οραναξίστες και οι προβλεπόμενες θαλάσσεις θα γίνουν και προσχώσεις που θα καταστρέψουν το Αττικό τοπίο στην ωραιότερη περιοχή ίσως του Σαρονικού. Παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, διότι πριν την κύρωση από τη Βουλή της Σύμβασης για το ελληνικό, ε, σταμάτησε η ανακήρυξη μεγάλου τμήματος του ελληνικού που είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν αρχαιολογικοί θησαυρία εκεί πέρα και επίσης παραβιάζεται η σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς για τους ίδιους λόγους. Τελειώνοντας, η ανάπτυξη που επιχειρείται στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι είναι γκρίζα και καταστροφή. Μιλά, συγγνώμη, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορούν οι μεταφραστοί να μεταφράζουν. Και τώρα ε, πρέπει να τελειώσετε γιατί περάσαμε με 8, 8 λεπτά τώρα. Τελειώνω. Σας έδωσα 5. Ε, να τελειώσω μια φράση. Ναι, ναι, βεβαίω. Ε, θεωρούμε ότι η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από μια πόλη 30.000 κατοίκων, αλλά ούτε μόλου, ούτε καζίνο, ούτε ουρανοξύστες Η περιοχή δηλώνω, σημειώνω ότι λέγεται ελληνικό. Η καταστροφή τη θεωρούμε ότι είναι μη αναστρέψιμη αυτή που προγραμματίζεται και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι ύβρις και νομοτελειακά ακολουθεί την έμεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Now, ε, we will Λοιπόν, να δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα περιβαλλοντικά ζητήματα πριν περάσουμε στον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες των αναφερόντων σήμερα και θα ήθελα να τους εγγυηθώ ότι συμμεριζόμαστε την άποψή τους σε σχέση με αυτό το ενδυνάμει σχέδιο. Θα ήθελα να διασαφηνίσω ορισμένα σημεία η περιβαλλοντική νομοθεσία ε, δεν ισχύει στην περίπτωση κύρωσης μιας σύμβασης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει τα σχέδια και προγράμματα αυτά που θα ε, ισχύουν ενδεχομένως στην ε, περιοχή του πρώην ελληνικού. Αυτό δυστυχώς εμπίπτει σε εθνικές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή όμως θα επαληθεύσει ώστε να ισχύσουν όλες οι περιβαλλοντικές ε, όλα τα περιβαλλοντικά προαπαιτούμενα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μία μελέτη αντικτύπου με βάση την οδηγία 2011 του 12 έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε μια τελική απόφαση. Δυνάμει αυτής της έρευνας θα γίνουν επαληθεύσεις και θα λάβουμε υπόψη και όλες τις άλλες ε, έρευνες. Θα λάβουμε υπόψη και την έρευνα στην οποία αναφερθήκατε εσείς και αυτό με βάση και τη μελέτη αντικτύπου. Εάν δούμε λοιπόν ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές της οδηγίας του 2012, τότε θα προβάλλουμε απαιτήσει. Υπάρχει αυτή η απέτηση για να δούμε κατά πόσο τα σχέδια αυτά μπορούν να ολοκληρωθούν με βάση την οδηγία 92 υπαριθμών 92. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας η οδηγία 2001-42 που αφορά τα περιβαλλοντικά δεν ισχύει. Οδηγία 2, του 2001-42 Ο νόμος 4062 ε, του 2012 μιλάει για εκτελεστικές πράξεις. Σε αυτή την περίπτωση θα δούμε ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και τότε οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να προβούν σε μια στρατηγική μελέτη. Σε σχέση με το περιβαλλοντικό σκέλος, παρακολουθούμε την εξέλιξη του σχεδίου και γι' αυτό οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τους αναφέροντες είναι ύψης της σημασίας. Επίσης, έχουν γίνει προσφυγές και ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα ζητήματα, γιατί ο εθνικός δικαστής θα πρέπει να εφαρμόσει το κοινοτικό δίκαιο. Δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Concerning the uh, για τις ενσυχίες για τις ε, κρατικές επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξεκαθαρίσει ότι σε ό,τι αφορά τον έλεγχο για τις κρατικές ε, επιδοτήσεις, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει το αν υπάρχει στρέβλος του διαγωνισμού ή αν υπάρχουν ωφέλη για συγκεκριμένες εταιρείε. Δεν είναι ο ρόλος της Κομισιόν να αξιολογήσει την σωστή ή λαθασμένη απόφαση μιας κυβέρνησης να πουλήσει, να εκμεταλλευτεί ένα χώρο. Ε, απλώς ελέγχει το, ε, αν τα κράτη-μέλη ε, στευλώνουν το, το, την ισότιμια όπλων ουσιαστικά μεταξύ των εταιριών στον ανταγωνισμό. Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μέτρα για τις κρατικές επιδοτήσεις πρέπει να, για, για αυτά τα μέτρα πρέπει να πληρούνται τέσσερι συγκεκριμένε προποθέσει. Για να υπάρχει κρατική επιδότηση, το μέτρο πρέπει να επηρεάζει τις, τους κρατικούς πόρους, πρέπει να δίνει ε, επιλεκτικό πλεονέκτημα σε κάποιες ε, εταιρείε και πρέπει να επηρεάζει τον ανταγωνισμό και το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Αν μία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρείται, τότε δεν έχουμε κρατική επιδότηση. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα. Σημειώνουμε ότι οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να πουλήσουν τη γη και τα οικήματα στο παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού, οργανώνοντας ένα διαγωνισμό το πούλησαν στη Lambda Development. Για την πώληση δεν λάβαμε οποιοδήποτε παράπονο, οποιαδήποτε καταγγελία και κανένας ανταγωνιστής δεν ε, παραπονέθηκε για το διαγωνισμό ή ότι έγινε κάποια ειδική παραχώρηση στην Lambda Developments. Δύο ερωτήματα βρέθηκαν για το θέμα αυτό το 2014 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ε, Μελετήσαμε το θέμα, το ερευνήσαμε, θέσαμε κάποια ερωτήματα στις ελληνικές αρχές δύο φορές, το 2014 και στις αρχές του 2015 και λάβαμε διευκρινήσεις από τις ελληνικές αρχές. Μετά τις οποίες το δικό μας το συμπέρασμα ήταν ότι δεν υπάρχει ανησυχία ούτε πραγματική ανάγκη να, να διερευνήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Γιατί η πώληση των ε, ε, οικημάτων ή του χώρου του ελληνικού μετά από διαγωνισμό ε, δίνεται στον, ε, ε, σε, όσον, σε όποιον, στον πλειοδότη και βεβαίω πρέπει να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ωφέλιμα για τον πλειοδότη. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, η Κομισιόν δεν έλαβε κανένα παράπονο, καμία καταγγελία των συμμετεχόντων ή των ανταγωνιστών ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο διαγωνισμό. Επίση, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει άλλο εξοδικαστικό ε, συμβασμό που μπορεί να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο. Οπότε τα πρακτικά θέματα που θα μπορούσαν να αποδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τον, με τον διαγωνισμό δεν υφίστανται. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να ε, διαρευνήσουμε περαιτέρω το θέμα. Επίσης, μιλήσατε για κάποια φορολογικά ωφελήματα, πλεονεκτήματα μετά την πώληση. Όντως, ζητήσαμε για το θέμα αυτό διευκρινήσεις από τις ελληνικές αρχές. Μας επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν ε, ε ελαφρύνσεις ε, για το ελληνικό ε, μετά την ιδιωτικοποίησή του και ούτε ειδική νομοθεσία ε, για τον, ε, η φορολογική ελάφρυνση για τον αγοραστή, για τη Lambda Developments. Οπότε δεν υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και εκπροσώπους των ελληνικών αρχών εδώ, ο κύριος Ορσοζίδης, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση. Έχετε το λόγο. Για το πολύ τέσσερα λεπτά. Τρία-τέσσερα λεπτάκια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Βρίσκομαι εδώ εκπροσωπούντα την ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα τον κύριο Σκουρλέτη, αρμόδιο υπουργό. Όσα ακούστηκαν ήταν πράγματι ενδιαφέροντα και από μέρου των ανθρώπων οι οποίοι αντιδρούν. Όλοι οραματιστήκαμε κάποια στιγμή ένα χώρο 6 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων σαν χώρο πρασίνου, όπου θα έδινε μια προοπτική ανάσταση στο λεκανοπέδιο. Τα χρόνια όμω τα οποία μπορούσε η Ελλάδα να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο πέρασαν ανεκμετάλλευτα και σήμερα βρισκόμαστε στα χρόνια τη κρίση. Υπό αυτέ τι συνθήκε λοιπόν ε, η προηγούμενη κυβέρνηση διαρρεύνησε τη δυνατότητα αξιοποίηση ή ε, ε, ιδιωτικοποίηση, όπω ακούστηκε, του συγκεκριμένου χώρου. Εμεί αναλάβαμε σαν κυβέρνηση τον Γενάρη του 2015. Το πρώτο μας μέλημα ήταν να εξετάσουμε τη σύμβαση, η οποία είχε ήδη υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και νομίζω ότι όλοι ομολογούν ότι την έχουμε βελτιστοποιήσει. Προσθέθηκε αντικείμενο ύψου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε έργα δημοσίου ενδιαφέροντο, τα οποία αφορούν στις υποδομές και δεν ήταν εξεκαθαρισμένο καθόλου στην προηγούμενη σύμβαση ότι αυτά ήταν ε, ε, υποχρέωση του, του αγοραστή. Συνεπώς το τίμημα συν 915 εκατομμύρια προσεγγίζει τα 2,5 δις. Όλα αυτά συνυπογράφησαν και εγκρίθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο, το αρμόδιο δικαστήριο το οποίο εγκρίνει τη συμβαση, δηλαδή ελέγχει κατά πόσο η σύμβαση στηρίζεται στη διακήρυξη ενό έργου. Από τη στιγμή που εγκρίθηκε από το ελεκτικό συνέδριο, νομίζω ότι όντω έχουν δίκιο τα μέλη τη Επιτροπή δεν συντρέχει λόγο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το διοικητικό μέρος. Σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό, η προσπάθεια που κατεβλήθη απέδωσε στο να διατηρηθεί περίπου το 51% της έκτασης, 2.600.000 τετραγωνικά μέτρα χώρος πρασίνου, απολύτως προσβάσιμος από όλους τους πολίτες, όπως και το παράκτιο μέτωπο, το οποίο πράγματι έχει 3.500 ε, μέτρα μήκος, εκ των οποίων το 1 χιλιόμετρο είναι η παραλία. Ε, θέλω να τονίσω ότι μέσα στις υποχρεώσεις του επενδυτή, οι οποίες προσθέθηκαν, είναι να αποθαρρύνει τους ε, πολίτες να προσεγγίζουν το χώρο με τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή, το μέσο σταθερής τροχιάς θα αναπτυχθεί σε, όλο, σε όλη αυτή την καινούργια πόλη που χτίζεται. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια επένδυση που θα φιλοξενήσει γύρω στους 27.000 ε, μόνιμους κατοίκους και άλλους 15.000 ε, εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, έγινε η προσπάθεια και άνοιξε όλο αυτό το πάρκο προς τους όμορους Δήμους, του Δήμου Ελληνικού, του Δήμου Αργιουπόλεως και του, ε, Δήμου ε, Είναι γνωστό επίσης ότι υπάρχουν αρχαιότητες στον υπόψη χώρο, όμως έχουμε μια αρχαιολογική υπηρεσία πάρα πολύ αυστηρή. Δεν είναι σωστό αυτό που γράφεται ότι μόνο 60 μέρες θα πρέπει να, να δίνεται λύση εφόσον προκύψουν αρχαιότητες ή να απομακρυνούνται. Με τη νέα τροποποιητική σύμβαση αυτό ο χρόνο είναι 110 ημέρε. Πρέπει δηλαδή να υποδείξει η αρχαιολογική υπηρεσία μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πώ θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα και υπάρχει μια ευελιξία που δεν πρέπει να ξεπερνά το 5% τη δομημένη επιφάνεια. Η δομημένη επιφάνεια, σύμφωνα με την καινούργια σύμβαση, δεν είναι 3.600.000 τετραγωνικά μέτρα, είναι 2.700.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό έγινε αποδεκτό, απλά το τονίζω και έχει συνυπογραφεί πλέον. Δεν λέω ότι είναι μικρή κλίμακα παρέμβαση, πράγματι είναι μεγάλη παρέμβαση, αλλά τηρηθήκανε κάποιες αναλογίες πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη και προτέρα κατάσταση. Οι αρχαιότητες λοιπόν προστατεύονται, υπάρχει αυτή η ελαστικότητα, μέχρι 5% από την προβλεπόμενη δομή στην επιφάνεια μπορεί να μειωθεί, χωρί να συντρέχουν λόγω καταγγελία τη σύμβαση και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Άλλωστε, ένα λόγο για τον οποίο οι επενδυτέ επέλεξαν την πατρίδα μου για να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο, δεν λέω ότι είναι ο μοναδικό, είναι πραγματικά το αρχαιολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Ελλάδα. Ούτε είναι τυχαίο ότι οι πρόγονοι <coughs> επέλεξαν να κατοικίζουν σε αυτόν τον τόπο. Πράγματι έχει όλα εκείνα τα προτερήματα τα οποία προσεγγίζουν. Με αυτόν τον τρόπο και με την επένδυση ολοκληρώνοντα, θέλω να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια να, να δικατηθούν ισορροπίες μεταξύ δομημένων και δομημένων του περιβάλλοντος, όσο είναι δυνατόν αυτό, και από την α, άποψη που δεν θα ήθελα να τη δεν είναι αυτός ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, αλλά είναι μια πραγματικότητα, θα δοθούν πραγματικά θέσεις εργασίας σε ανθρώπους που κυριολεκτικά υποφέρουν στην πατρίδα μου αυτήν την χρονική περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να ακούσουμε τα μέλη. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι εδώ αγαπητοί συνάδελφοι με διπλή ιδιότητα. Πρώτον, είμαι άμεσα ενδιαφερόμενος για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης διότι αν μεγιστοποιηθεί λιγάκι ο χάρτης του ελληνικού, δίπλα θα δω το σπίτι μου. Δεύτερο, και επομένω τις ανησυχίες τις ζω και θα τις βιώσω ευθέως. Δεύτερο, ως ε, Έλληνας βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας αυτής γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πρόβλημα, γνωρίζω το μέτωπο που είχε υπάρξει και υπάρχει Δυστυχώ υπήρξε επαναχώρηση τη κυβέρνηση σχετικά να μην προχωρήσει αυτή η εκποίηση. Τρίτο, ω Ευρωβουλευτή που δεν είμαι τώρα μέλο τη Επιτροπή Αναφορών, αλλά ήμουν στο παρελθόν μέλο τη Επιτροπή Αναφορών για να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει τη θετικότερη γνώμη στο ελληνικό κοινό, διότι οι αναφορές που έθηκαν τα προβλήματά του αντιμετωπίστηκαν με την απαραίτητη ευαισθησία δεν θεωρώ ότι θα είμαι χρήσιμος αν επαναλάβω τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα της, ε, της Επιτροπής Αναφορών για παραβιάσεις τόσο της ε, συνθήκης λειτουργίας όσο και τις παραβιάσεις όλου, θα έλεγε κανείς, του διεθνούς ευρωπαϊκού πρωτογενούς και δευτερογενούς κόρπους όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος. Απλώς θέλω σύντομα να σχολιάσω κάποιες απαντήσεις που δόθηκαν από την πλευρά της Κομισιόν και από τον συνάδελφο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κομισιόν, δεν είναι ακριβές αυτό που λέγεται, ότι ο νόμος αυτό δεν υπάγεται και δεν πρέπει να υπακούει, ο νόμο 40, να υπακούει στην οδηγία εκεί. Υπάρχει μια μακρά ιστορία, αυτό ο νόμος έγινε κατά παραβίαση τη πάγια χωροταξική ε, ρύθμιση, για να ξεφύγει η δυσκολία αυτή από μια παλιά ρύθμιση που απαιτούσε και σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε παραβίαση διότι δεν λήφθη υπόψη η απέτηση για στρατηγική ε, σχεδιασμό περιβαλλοντική επίπτωση. Δεύτερον, η παραπομπή της Κομισιόν ότι είναι ορισμένα ζητήματα που πρέπει κανείς να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη. Επειδή έχω προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη μαζί με άλλους, σας λέω αγαπητοί συνάδελφοι, ότι όταν ισχυρίζονται οι αναφέροντες ότι έχει παραδιαστεί η Διεθνή Συνθήκη του Άρχους, μιλάμε και για τους τρεις πυλώνες, και για την πληροφόρηση, και για τη συμμετοχή και για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, έχει φτιαχτεί έτσι ο νόμος, έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του εποπτικού συμβουλίου που παραπέμπεται αυτή η υπόθεση, ούτω ώστε να μην μπορείς να πας εκεί. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορείς να παραπέμπεις το θέμα εκεί. Για αυτούς που λένε ότι η ελληνική δικαιοσύνη τα κρίνει. Δεν τις έχουν κόψει τα φτερά, τις έχουν αποτρέψει αυτή τη δυνατότητα. Τέλος, ε, αυτό που ήθελα να σας πω όσο αφορά το που είπε η εκπρόσωπος που μίλησε για τον ανταγωνισμό και τις κρατικέ ενισχύσεις. Όντω. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα δεν υπήρχε άλλος στο διαγωνισμό, υπήρχε ένας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν παραβιάσεις τόσο στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσο και στον ανταγωνισμό με τη γενικότερη έννοια. Έχουμε ένα προηγούμενο στην Ελλάδα με μια εκποίηση του λιμανιού στην Κόσκο όπου επισημάνθηκαν και με δικέ μου ερωτήσει και άλλε, έγιναν φοροαπαλλαγέ εκτεταμένε και ήρθε μετά από τρία χρόνια η Κομισιόν να αναγνωρίσει ότι όντω είχαν γίνει αυτέ οι παραβιάσει. Καταλήγω λοιπόν, με συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει παραδεκτή η αίτηση ε, των αναφορών ε, και θα πρότεινα εκ τη εμπειρία που έχω για να πάρουμε επίσημη απάντηση σε αυτά τα θέματα γιατί θεωρώ ότι πρέπει η Επιτροπή να βασανιστεί πολύ σε αυτά τα ζητήματα να καταθέσει η Επιτροπή σας δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς μπορώ να το κάνω μεμονωμένα, προφορική ερώτηση προ την Κομισιόν με το θέμα αυτό, για να γίνει και με συζήτηση, να προετοιμαστεί καλύτερα η Κομισιόν στι απαντήσει που σήμερα μα δόθηκαν, για να πάρουμε μια απάντηση αν όντω ισχύουν, εγώ λέω ισχύουν, οι ενστάσει τη Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τον χρόνο που μου διαθέτετε. Ευχαριστώ, κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα επισημάνω κι εγώ αυτό που είπατε προηγουμένως, ξεκινώντας, ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά και ταυτόχρονα απίθανο να εκπροσωπεί ένας βουλευτής την κυβέρνηση ενός κράτους. Διότι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι διαφορετικό όργανο από την νομοθετική εξουσία. Και είναι προφανές ότι σε αυτήν εδώ την Επιτροπή το Υπουργείο μπορεί να το εκπροσωπήσει ο Υπουργό, ο Υφυπουργό, ο Γενικό Γραμματέα, η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Είναι ιδιαίτερα παράδοξο να υπάρχει εξουσιοδότηση της κυβέρνησης για εκπροσώπησή του από ένα βουλευτή. Δεν αφορά βέβαια εσάς εδώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι και αντισυνταγματικό. Διότι δεν μπορεί ένα βουλευτή εκ τη ιδιότητό του να εκπροσωπείται η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό παραβιάζει την αρχή τη διάκριση των εξουσιών στην Ελλάδα. Αλλά δεν αφορά τη δικιά σα επιτροπή. Είναι πάντως παράδοξο για την δεύτερη φορά που η ελληνική κυβέρνηση δεν εμφανίζεται στην επιτροπή αυτή. Είχε κληθεί και στο θέμα των οφειλών, των γερμανικών οφειλών με την επιστολή που είχατε αποστείλει και τελικά εμφανίστηκε εδώ πάλι η ελληνική κυβέρνηση μέσω Ευρωβουλευτή που μετέφερε το μήνυμα του Προέδρου της Βουλής ο οποίος μας έλεγε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα τι έχουμε εδώ στο θέμα. Θα πάω στο κομμάτι πρώτα απ' όλα των κρατικών ενισχύσεων. Είπε η Κομισιόν ότι επειδή είχαν γίνει δύο ερωτήσεις το έτος 2014, εξέτασε την υπόθεση και είδε ότι δεν υπάρχουν βασικά προβλήματα. Να ενημερώσουμε την Κομισιόν ότι υπάρχει καινούριο νόμος, ο οποίος οριστικοποίησε την μεταβίβαση της, α, ε, ε, του ελληνικού ΑΕ στην συγκεκριμένη εταιρεία στη Lambda Development. Και ρωτώ εγώ την Κομισιόν, αν είναι ή δεν είναι κρατική ενίσχυση το εξή. Προκειμένου να γίνει μεταβίβαση ε, ακινήτων στην Ελλάδα, πληρώνει κανείς φόρο τη προστιθέμενης αξίας 23%, ίσως και 24%, πληρώνει φόρο μεταβίβασης 11% και πληρώνει και φόρο υπεραξίας. Ο νόμος λοιπόν 3943 του 2011 απαλλάσσει την εταιρεία ελληνικών ΑΕ, άρα και την, ε, τους, αυτούς τους επενδυτές σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών που αγόρασαν την εταιρεία, από τι? Από κάθε φόρο, αμοιβή, που συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος για κάθε μορφή εισόδημα που προκύπτει, από φόρο μεταβίβασης, από φόρο συγκέντρωση κεφαλαίου, από φόρο έναρξης δραστηριοτήτων, από τέλος εισφοράς δικαιώματος υπέρ του δημοσίου, από τέλος υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών και αμοιβών συμβολιογράφων, δικηγόρων κλπ. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα ένα μεγάλο πρόβλημα κατά τη μεταβίβαση ακινήτων είναι ότι πληρώνεις όλα αυτά και εν προκειμένου εδώ δεν υπάρχει καμία πληρωμή. Υπάρχει απαλλαγή όλων των φόρων. Αυτό δεν είναι καραμπινάτη κρατική ενίσχυση. Τι σημαίνει πρακτικά κρατική ενίσχυση. Δεύτερον, ο νόμος ο οποίος ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, ένας νόμος του 1953, ο οποίος έχει εισαχθεί μάλιστα και με συνταγματική ισχύ στην Ελλάδα, ε, δίνει δυνατότητα φοροαπαλλαγών και αυτός ο νόμος είναι νόμος στον οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη μεταβίβαση. Είναι ο νόμος 2687 του 1953 και εκεί προβλέπει απαλλαγές, φόρο Εδώ έχετε μια περίπτωση αντίστοιχη με αυτή της Ιρλανδίας, όπου εκεί υπήρχαν τεράστιες φοροαπαλλαγές, στην περίπτωση της Apple. Άρα λοιπόν δέστε τα θέματα ξανά, διότι είναι ξεκάθαρες οι περιπτώσεις της παραβίας αυτής. Δεύτερον, Έχω υποβάλει ερώτηση στην Κομισιόν στις 28 Μαΐου για το θέμα του ελληνικού. Αναφερόμουν στο άρθρο 107 για τις κρατικές ενισχύσεις. Μου απήντησε ο κύριος Βέλα εν προκειμένο ότι εάν οι εθνικές αρχές θεωρούν ότι υπάρχει ε, κρατική ενίσχυση, να ενημερώσουν την Κομισιόν. Απίθανα πράγματα. Όταν σας έκανα εγώ την ερώτηση, σας την έκανα για να διερευνήσετε εσείς αν υπάρχει κρατική ενίσχυση. Δεν θα σας πει το κράτος αν έχει κάνει κρατική ενίσχυση. Δεύτερον, έχετε πλέον την αναφορά η οποία το καταγγέλει. Άρα λοιπόν έχετε επίσης οψιγενές γεγονός. Ποιο? Ότι τώρα μόλις ψηφίστηκε ο νόμος για την παραχώρηση. Άρα λοιπόν πρέπει να εξετάσετε το θέμα αυτό. Έρχομαι, σύντομα κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Έρχομαι στο θέμα των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Έθετα αυτά τα θέματα στην ερώτησή μου. Και η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Βέλα είναι εν προκειμένου πολύ συγκεκριμένη και δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει ή αν επικοινωνεί η μία, η μια επιτρο... διεύθυνση επιτροπής με την άλλη. Διότι αναφέρεται εν προκειμένου στην υποχρέωση και αυτά είναι αντίθετα από αυτά που μας είπαν. Λέει λοιπόν ότι όλες οι απαιτήσει της οδηγίας 2001, τις απαιτήσει 92-43 πρέπει όλες αυτές οι απαιτήσει να υπάρχουν και να τηρηθούν πριν την έγκριση του έργου. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Δέχομαι αυτό που είπατε εσείς της Κομισιόν ότι πρέπει να πάτε να τα δείτε από κοντά. Και είμαι σύμφωνος ότι πρέπει πλέον να γίνει επιτόπου έλεγχος. Προτείνω λοιπόν τα εξή. Πρώτον, να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά. Δεύτερον, να γίνει μεταβασή της ίδιας της Κομισιόν επιτόπου και φυσικά αν θέλετε και τη επιτροπή Αναφορών σε μια fact-finding mission για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει. εμεί ξέρουμε, αλλά να δουν οι υπόλοιποι και να δει και η Κομισιόν. Τρίτον, να λάβει υπόψη η, η Κομισιόν τα όσα τις αναφέρουμε σήμερα περί κρατικών ενισχύσεων και φοροαπαλλαγών, να ζητήσει διευκρινήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Εδώ κυρία Πρόεδρε πρόκειται για μια υπόθεση την οποία έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως διότι πρόκειται για μια παραχώρηση, υποχρέωση που έχουν επιβάλει οι δανειστές στην Ελλάδα η υπάρχουσα κυβέρνηση ήταν στις πολιτικές δυνάμεις που μαζί μας και με τους υπόλοιπους συναδέλφους είχαμε αντιταχθεί σε αυτή την παραχώρηση του ελληνικού τώρα εφαρμόζει την, το, την παραχώρηση αυτή διότι είναι στα προαπαιτούμενα. Προκειμένου να πάρει τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν τα πήρε, πέρασε τη ρύθμιση αυτή τελευταία στιγμή από την Ελληνική Βουλή. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία επιβολή εκ μέρους των δανειστών στην υπόθεση του ελληνικού παραχώρησης δημόσιας περιουσίας η οποία έχει πολύ σημαντική αξία και η οποία φυσικά δεν ανταποκρίνεται η μεταβίβασή της στο τίμημα το οποίο έχει δοθεί. Υπάρχουν όμως όλες οι παραβιάσεις που σας αναφέραμε και θέλουμε να εκτιμηθούν από την Κομισιόν. Να παραμείνει λοιπόν ανοιχτή η υπόθεση αυτή και να την ξανασυζητήσουμε εδώ όταν θα έχουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα ο λόγος είναι για κυρία Σακοράφα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα σας καλούσα, κυρία Πρόεδρε, όπως και τους συναδέλφους και όποιον βρίσκεται μέσα σε αυτή την αίθουσα, να κοιτάξετε καλά αυτή την περιοχή και να δείτε ότι είναι η πιο ακριβή περιοχή της Αττικής. Η πιο ακριβή περιοχή της Αττικής. Ο επιχειρηματίας που αγοράζει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα, αγοράζει με λιγότερο από 100 ευρώ το τετραγωνικό, όταν το ίδιο το δημόσιο αγοράζει δίπλα με 2,5 και 3 χιλιάρικα το τετραγωνικό. Αυτό είναι το ένα και απορώ πώς έρχεται ο κύριος Σουζουνίδη σήμερα σε αυτή την Επιτροπή εκπροσωπώντας μια αριστερή κυβέρνηση να υπερασπιστεί όσα υπερασπίστηκε προηγουμένως. Να υπερασπιστεί την πιο σκληρή απικιακού τύπου σύμβαση που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση. Πραγματικά απορώ. Θα σας αναφέρω μόνο ένα γιατί εδώ δεν είναι θέμα του πώς τσακωνόμαστε εμείς στην Ελλάδα σε σχέση με τα εσωτερικά μας τα πολιτικά, αλλά μέσα από τη σύμβαση και θα σας στείλω σε όλους κύριοι συνάδελφοι τα στοιχεία της σύμβασης, θα σας διαβάσω μόνο ένα σημείο που λέει ότι έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες θα πρέπει να απορρίπτουν όλες τις ασκηθήσεις αιτήσεις ακυρώσεως, είναι αιτία ανέρεσης της σύμβασης. Το καταλαβαίνετε αυτό αν τολμήσει το ανώτατο δικαστηρίο να βγάλει μια απόφαση αναιρετική, η σύμβαση θα καταπέσει και το ελληνικό δημόσιο, στον κύριο επιχειρηματία, τον οποίο ευνοεί αυτή η κυβέρνηση, θα πρέπει να πληρώσει τόσα και άλλα τόσα από όσα πλήρωσε. Δεν θα αναφερθώ σε όσα αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, για να μην σα κουράσω. Αυτό που θέλω να πω όμω ότι η αναφορά που συζητάμε σήμερα έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από Έλληνε πολίτε που αγωνιούν και αγωνίζονται πραγματικά για τη διάσωση του περιβάλλοντο αλλά και τη δημόσια περιουσία στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή εξαφανίζεται και που είναι το μόνο πράγμα που έχουμε στα χέρια μα αν μπορούμε κάποια στιγμή και θέλουμε να βγούμε από την κρίση που βρισκόμαστε. Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν καταθέσει πάρα πολλοί πολίτε ε, ε, στο δικαστήριο και στους, ε, στη, στη δικαιοσύνη αναφορές και μηνύσεις. Πάρα, πολιτική, πάρα πολλοί πολιτικοί μεταξύ των οποίων και εγώ έχουν κάνει αναφορές και δεν έχει να κάνει με πολιτικό φορέα, είναι από διάφορους πολιτικούς φορείς και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι για μας κυρία Πρόεδρε να καταφέρουμε να μετατρέψουμε αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση με τρόπο τέτοιο ώστε τελικά να αποβεί προ όφελο των κατοίκων της πόλης, της χώρας και κατ' επέκταση γιατί αυτή η έκταση είναι ένα τεράστιο έργο για την Ελλάδα. Θα πάω σε αυτά που αναφέρθηκε η Επιτροπή εν συντομία. Στην, στην, παραβίαση και αν υπάρχει της συνθήκης άρχους. Υπάρχει παραβίαση της συνθήκης άρχους καθότι δεν έγινε ποτέ, κυρία Πρόεδρε, δημόσια διαβούλευση και δεν γνωρίζω η Επιτροπή που στηρίζεται και απαντά ότι δεν έχει γίνει παραβίαση. Το συγκεκριμένο θέμα το παρακολουθώ πάρα πολύ κοντά από την αρχή της εξαγγελίας της ελληνικής κυβέρνησης για τη δίθεν αξιοποίηση του ελληνικού και σας διαβεβαιώ προσωπικά ότι τέτοιου είδους διαβουλεύσεις δεν έχουν γίνει ποτέ, ούτε φυσικά ποτέ έχει συνεκτιμηθεί η άποψη των κατοίκων, οι οποίοι δίκαια αγωνιούν για την περιβαλλοντική καταστροφή της περιοχής, μιας περιοχής που θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελευταίο πνεύμα οξυγόνου της Αθήνας. Όσον αφορά τα μεμονωμένα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν και που πρέπει να, να, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες 2011-92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να, να παρακολουθεί η Επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, αν τελικά παραβιάζονται αυτές οι οδηγίες. Στις περιβαλλοντικές μελέτες. Στην αναφορά επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικής εκτίμησης βάσει της οδηγίας 2001 κάθετο 42 και για την οποία η Επιτροπή μας ενημερώνει ότι επειδή δεν έχουν εγκριθεί οι κανονιστικές πράξεις, δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της σχετικής οδηγίας. Δεν πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να το παρακολουθήσει ώστε να διαπιστώσει αν παραβιάζεται η οδηγία ή όχι. Σε παρόμοια θέση θα αναφέρω πάλι και επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε και συγγνώμη αν μιλάμε περισσότερα από όσο πρέπει αλλά μα καίει αυτό το θέμα. Σε παρόμοιο θέμα πριν από 15 χρόνια, με τον ίδιο, προσέξτε, με τον ίδιο επενδυτή, το τονίζω αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, και την ίδια τακτική που ακολούθησε στα θέματα της διαδικασία, τη επένδυσής του, στο Μαρούσι όταν ήμουν δημοτική σύμβουλος, ανοιγέται ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο που κατέστρεψε την, την περιοχή και οικιστικά και οικονομικά, αν θέλετε αυτό χαρακτηρίστηκε το μεγαλύτερο ευθέρετο της Ευρώπης και από πρώην Πρωθυπουργού και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο αυτό της χώρας μας, το έκρινε καταδευστέο και παράνομο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ξέρετε τι κάνει. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, αυτό το συγκεκριμένο που το Συμβούλιο της Επικρατείας το έχει ε, ε, ε, χαρακτηρίσει παράνομο και πρέπει να καταδαφιστεί, να βρει έναν τρόπο να το διασώσει, να μην πληρώσει πρόστιμα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εάν αυτή η Επιτροπή κάποια στιγμή δεν αποφασίσει που λειτουργεί, που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ε, να, να, να προσπαθήσει να προστατεύσει αυτού του είδους της περιουσίας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την, το, το αν, υπάρχει, αν υπάρχουν ε, στους όρους ανταγωνισμούς ε, που αναφέρθηκε από τους άλλους συναδέλφους, δεν θέλω να, να, να απαντήσω πάνω σε αυτά. Υπάρχουν ξένα δημοσιεύματα που θα ε, που ήθελαν, πραγματικά ήθελαν εταιρείε με πολλαπλάσιο τίμημα να συμμετάσχουν στην, στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ε, ε, και είδαμε που κατέληξε. Είναι ένας ο, ο επενδυτής, υπάρχουν ε, δημοσιεύματα από ξένες εφημερίδες, από πολύ μεγάλες εφημερίδες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, έχει κάνει έρευνα η Επιτροπή αν τηρήθηκαν οι αρχές του ανταγωνισμού που επιβάλλει η Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, στην, στην μέσα στην αγορά τη Έχουν γίνει όλα αυτά. Γιατί δεν άκουσα τίποτα για, για αυτά να μας λέει η Επιτροπή. Και κλείνω κυρία Πρόεδρε, για, ε, που να, να, απαντήσω για την, να, να αναφερθώ στην παραβίαση του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Επιτροπή μας ενημερώνει ότι μετά από ερωτήσεις προς τις ελληνικές αρχές δεν διακρίνει παραπέρα λόγους διερεύνηση των ισχυρισμών των αναφερομένων. Πιστεύω ότι η Επιτροπή θα έπρεπε παραπέρα να διαρευνήσει αυτό το θέμα, καθώς η απάντησή της νομίζω ότι προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Στην Ελλάδα ξέρουμε όλοι ότι η Σύμβαση του Ελληνικού είναι το απάβγασμα της διαπλοκής και του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και μάλιστα μιας περιουσίας που πουλιέται αντί πινακίου φακής. Μετά από όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε και κυρία συνάδελφε, δεν νομίζω ότι μια τέτοια αναφορά πρέπει να, παρα... να... θα πρέπει να κλείσει, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ε, για παραπέρα διαρεύνηση φυσικά, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, την σοβαρότητα και το κύρος που έχει αυτή η Επιτροπή. Θα πρέπει, πιστεύω, να γίνει μια επιτόπια επίσκεψη για να δείτε πραγματικά και εσείς από κοντά την πραγματικότητα που εμείς προσπαθούμε εδώ να σας περιγράψουμε και να, να σας χαρακτηρίσουμε. Και φυσικά, κυρία Πρόεδρε, θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνει μια προφορική ερώτηση και συζήτηση στην Ολομέλεια για το ελληνικό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και για όλες τις ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ και δεν, δεν βαριέμαι ποτέ όταν μιλάει ο άνθρωπος με πολύ πάθος, όπως μιλήσατε εσείς τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα είναι ο λόγος για τον κύριο Κύρκος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να συμφωνήσω και εγώ με τις επισημάνσεις του συναδέλφου του κυρίου Μαριά για την εκπροσώπηση της ελληνικής κυβέρνησης. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι καταλαβαίνουμε πως το έργο του εκλεκτού συναδέλφου του κυρίου Ρουσουζίδη ήταν σήμερα να διαλύσει κάποια όνειρα, οπότε συμπάσχοντας αυτό το δύσκολο ομολογουμένο έργο δεν θέλω να του φορτώσω κι άλλο βάρος τι γίνεται στο ελληνικό. Είναι πραγματικά, όπως είπε η κυρία Σακοράφα, ένα από τα πιο σημαντικά, πιο ακριβά οικόπεδα στο χώρο της Αττικής. Όμως 15 χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις οραματιζόντουσαν επενδύσεις στα λόγια και στην πράξη έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο και δυστυχώς φιλοξενεί και μερικές χιλιάδες προσφύγων σε συνθήκες που δεν είναι, δεν προσφέρουν αξιοπρεπή διαβίωση. Σε αυτά τα 15 χρόνια η σημερινή κυβέρνηση, κόμμα της αντιπολίτευσης, το έκανε όχι απλώς είχε μια πολιτική αντίθεση στη συγκεκριμένη επένδυση, αλλά όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός μας είχε πει, είναι η σημαία του αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, του δημόσιου χώρου. Μια τέτοια σημαία η οποία με, την, ε, με το ρεαλισμό που απαιτείται από μια κυβέρνηση όταν έρθει στην εξουσία βλέπουμε ότι κατεστάλλει αυτή η σημαία και βεβαίως οι πολίτες οι οποίοι, τόσα χρόνια στήριξαν μια τέτοια προσπάθεια νιώθουν και είναι σίγουρο ότι νιώθουν προδομένοι. Υπεστάλλει, σωστά. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Η προσπάθεια της κυβέρνησης δεν κατεστάλλει διότι μπορεί να ήρθε στην Ελληνική Βουλή και να πλησφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία εκτός από δύο κόμματα το σημερινό σχέδιο, όμως μέχρι να φτάσει στη Βουλή είχαμε δει παρεμβάσεις των Υπουργών, αν θυμηθούμε παλιότερα τις αναπληρώτερες Υπουργού Οικονομικών που είχε δώσει ένα κομμάτι για να ε, γίνεται διαχείριση των, αποβλήμα, των απορρίτων, των απορριμμάτων, ο Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντο, ο οποίο δήλωσε ότι η επένδυση θα απαξιωθεί από την αγορά, και ο Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίο θέλησε να βάλει κάθε ε, διοικητική πράξη κάτω από τον έλεγχο της αρχαιολογικής υπηρεσίας ώστε να μην εκδοθεί ποτέ κανένα, ε, κανένα σχέδιο. Αυτά τελικά η κυβέρνηση κατάφερε και τα ξεπέρασε ε, και προχωρήσαμε στην ψήφιση στο Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, τις δυνατότητε να γίνει επένδυση. Τώρα, επειδή δεν θέλω μόνο να διαλύουμε όνειρα, αλλά θέλω να βάζω και όνειρα, για μένα όνειρο θα ήταν πραγματικά η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με έναν τρόπο που να μπορέσει να προκαλέσει επενδύσεις μικρές ή μεγάλες, να φέρει θέσεις εργασίας, μικρέ η ανεργία παρά μόνο με ιδιωτικές επενδύσεις. Δυστυχώς οποιοδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλος τρόπος κρατικής παρέμβασης ανήκει στα όνειρα τα οποία αναφέραμε πριν. Μπορούμε λοιπόν να φερει θέσει εργασιας γιατι δεν υπαρχει κανενας αλλος τροπος να μειωθει η ανεργια παρα μονο με ιδιωτικέ επενδυσεις δυστυχώ, οποιοδηποτε αλλο αλλος τροπος κρατικης παρεμβασης ανηκει στα ονειρα τα οποια αναφεραμε πριν μπορουμε λοιπον να δουμε τους όρους κάτω από τους οποίους αυτές οι επενδύσεις και με την παρέμβαση και και συμμετοχή των πολιτών, όπως είναι οι πολίτες που έρχονται σήμερα και κάνουν την αναφορά, να εξασφαλίσουμε πως, ας πούμε, για το Β και το Ε που αναφέρεται στην, ε, στην περίληψη που μας δώσατε, για τις λεπτομέρειες δηλαδή που δεν γνωρίζει ο κόσμος, ξέρουν πως εκκρεμεί ακόμα το master plan. Δεν έχει δημοσιευθεί. Δεν έχει ε, εγκριθεί από την περιφέρεια Αττικής. Δεν έχει οθετηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι ένας ε, αγώνας ο οποίος πρέπει να δοθεί ώστε να μην μπορέσει τίποτα το οποίο είναι έξω από τον νόμο να περάσει. Είναι ένας δρόμος λοιπόν που έχει να ακολουθηθεί. Τώρα για τα λιβάδια της Ποσειδονίας, τα φύκια δηλαδή του βυθού ή τον κίνδυνο των ακτών από τη δόμηση, δεν έχω δει σε κανένα μέρος του σχεδίου να αναφέρεται παρέμβαση στην ακτή ή το βυθό. Άρα θα έλεγα πως είναι ε, πολύ ενδιαφέρουσα ε, η το βυθο αρα θα ελεγα που ειναι πολυ ενδιαφερουσα η παρεμβαση για την προστασία αυτών των περιοχών. Όταν κινδυνεύσουν πραγματικά πρέπει να τις προστατεύσουμε, αλλά προς το παρόν δεν βλέπουμε τέτοιο έργο. Ποια είναι η ουσία αυτών των πραγμάτων. Η ουσία είναι ότι για να έχουμε επενδύσει πρέπει να έχουμε φορολογικό περιβάλλον σταθερό, πολιτική σταθερότητα και η διοικητική ικανότητα να τη φέρουμε εις πέρας. Το πρώτο δεν το έχουμε, το δεύτερο κατά ένα μέρος το έχουμε αλλά και δεν το έχουμε, το τρίτο σίγουρα δεν το έχουμε και είναι αυτό στο οποίο πρέπει οι Έλληνες πολίτες να δώσουν τη μάχη. Ούτε να μπορούν να ξεπεραστούν οι διοικητικές αδυναμίες προς όφελος ανεξέλεγκτων πράξεων του επενδυτή, ούτε φυσικά από μόνες τους να αποτελέσουν ένα βραχνά ώστε να μην μπορέσει να υλοποιηθεί η ε, επένδυση. Για το θέμα, και κλείνω με αυτό, για το θέμα του τιμήματος, το οποίο ε, μέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν ελάχιστο και ξαφνικά φάνηκε πως είναι μεγάλο και ε, έρχεται σε, ε, ας πούμε, δίνει τη σωστή αξία της επένδυσης, μπορώ να πω πως το μέγεθο μια επένδυση εξαρτάται από το ενδιαφέρον που δείχνουν και άλλοι επενδυτέ να συνεισφέρουν. Βλέπουμε πω η συγκεκριμένη επένδυση έγινε από μία μόνο εταιρεία και ξέρουμε πολύ καλά ότι τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για τη γη είναι ένα μικρό μέρο των χρημάτων που συνολικά θα επενδυθούν ώστε να μπορέσει αυτός ο χώρος να αποδώσει για τον επενδυτή αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει και στο κοινωνικό σύνολο είτε μέσω του φορολογίας είτε μέσω των θέσεων εργασίας που θα ε, υλοποιηθούν. Άρα οι πολίτες πρέπει να επαγρυπνούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από εδώ και πέρα, αλλά να συγκεντρωνόμαστε και σε αυτό που είναι εφικτό να γίνει και όχι μόνο σε αυτό που ονειρευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ξαφνικά έγινε η Επιτροπή μας ελληνική. Τι να κάνουμε, αλλά τώρα είναι... Μέχρι πρόσφατα ήταν ισπανική για αρκετέ φορέ Επομένω. Ισπανική, αλλά τώρα, τώρα έχουμε μια συνάδελφη από, από την Γερμανία. Και τώρα θα, θα, I, would, now give the floor to you, Ska. Να δώσω το λόγο σε σένα, Ska. Αναζωογονητικό. Να έχουμε Ελληνική Επιτροπή μένα, αλλά και Ευρωπαϊκή ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι μιλάς ε, ελληνικά, Σεσίλια. Ευχαριστώ τους αναφέροντες που είναι παρόντες σήμερα, που έκαναν όλη αυτή την προσπάθεια και τη δουλειά για το θέμα αυτό και από εμάς, από τους Πρασίνους. Ε, όντως δημιουργούνται πολλές ανησυχίες, ε, πολλά από όσα μας ανησυχούν και εμάς ήδη έχουν αναφερθεί, αλλά για να μπω λίγο σε λεπτομέρειες για τα θέματα τα περιβαλλοντικά. Μία από τις βασικές μας ανησυχίες είναι ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Περιβάλλον και δεν χρειάζεται να σας πω όλες τις οδηγίες, θα πρέπει να υπάρχει ε, αξιολόγηση δικτύπου περιβαλλοντικού που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Ε, βλέποντας και την περιοχή, βλέποντας και τα περιβαλλοντικά ενδιατήματα που περιλαμβάνονται, ας πούμε τα λιβάδια Ποσειδονίας, που είναι ένα είδος φυκιού αν δεν το ξέρετε, νομίζω ότι είναι σημαντικό ένα μια τέτοια στρατηγική ε, αξιολόγηση δικτύπου, περιβαλλοντικού δικτύπου πρέπει να γίνει, σύμφωνα και με την νομοθεσία, την ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη, επαρκώς τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς το παρόν αν κατάλαβα καλά, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή τη είπε ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμή, άρα δεν έχει υπάρξει παραβίαση. Ε, ναι, αλλά αν ε, δούμε τα πράγματα αυτή τη στιγμή έχει γίνει η ζημία, δεν κάνουμε τίποτα. Το θέμα είναι τη αξιολόγηση αντικτύπου να γίνει πριν γίνει η καταστροφή στο περιβάλλον. Αν ε, η καταστροφή γίνει πρώτα και μετά κάνουμε την αξιολόγηση αντικτύπου, δεν μπορούμε να διορθώσουμε τη ζημιά, ούτε μπορούμε να ξαναφέρουμε πίσω σύντομα τα λιβάδια Ποσειδονία, αν τα αφήσουμε πρώτα να καταστροφούν. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η λάθο προσέγγιση να κατόπιν ορτής να στεναχωριόμαστε. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι αυτή η συγκεκριμένη περιοχή δεν προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000. Αλλά αυτό ήδη μπορεί να είναι πρόβλημα από μόνο του. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτή είναι ακριβώ μια περιοχή που θα έπρεπε να εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000. Οπότε αναρωτιέμαι, μήπω η Κομισιόν θα έπρεπε να κοιτάξει περισσότερο το θέμα των εθνικών υποχρεώσεων που έχουν να κάνουν με, την, ε, με το χαρακτηρισμό ε, περιοχών ε, Natura 2000 και κατά πόσο αυτές πληρούνται. Το Natura 2000 δεν το βρήκαμε, δεν το εφήβραμε χτες. Είναι ένα θέμα νομίζω που θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί. Οπότε, αν η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν είναι 2000, περιοχή Natura 2000, άρα δεν χρειάζεται συγκεκριμένη προστασία, νομίζω ότι δεν του δίνεται ιδέουσα προσοχή. Θα έπρεπε η περιοχή να είναι Natura 2000, αλλά δεν έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί λοιπόν η νομοθεσία σχετικά για μια, όπως, θα γινόταν για μια, όπως θα γινόταν για μια περιοχή Natura 2000. Βεβαίω είναι σημαντικό να εμπλακεί και η τοπική κοινωνία στον ε, σχεδιασμό. Οι συνάδελφοι το είπαν ήδη αυτό. Τώρα για τις κρατικές επιδοτήσεις για τις κρατικές ενισχύσεις να επιστήσω την προσοχή της Κομισιόν σε μια ε, υπόθεση ε, της ε, Κομισιόν για την, με τη Γαλλία για μια εταιρεία ναυτιλιακή όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αν υπάρχει μόνο ένας στο διαγωνισμό που πληρεί τα κριτήρια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κρατική επιδότηση επειδή υπάρχει διαδικασία διαγωνισμού. Βλέποντας λοιπόν αυτή την περίπτωση της Γαλλίας δεν ξέρω κατά πόσο η επιχειρηματολογία σας ε, όντως μπορεί να ισχύει πάντα. Οπότε εμείς ως πράσινοι ζητούμε η αναφορά αυτή να μείνει ανοιχτή και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περαιτέρω ενημέρωση για το κατά πόσο η περιοχή αυτή που έχει τα ε, λιβάδια Ποσειδονίας θα έπρεπε να ενταχθεί στην Natura 2000. Γιατί ε, υποτίθεται ότι στο χώρο εκεί θα δημιουργηθεί και μαρίνα, που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων θα υπάρξει ζημιά στα λιβάδια Ποσειδονία. Και επίση είναι, ενδιαφέρουσα η υπόθεση αυτή, γιατί το θέμα αυτό των ιδιωτικοποιήσεων είναι όντω σημαντικό και είναι κομμάτι του πακέτου. Βλέπουμε λοιπόν να ζητούμε την, από την Κομισιόν να δει μία αναφορά από την μία λέμε στην Ελλάδα ιδιωτικοποιήστε αυτή την περιοχή και από την άλλη λέμε στην Κομισιόν α, δείτε λίγο την ιδιωτικοποίηση που έγινε στην Ελλάδα. Μήπως πρέπει να ζητήσουμε να αναθερωθεί ή να, να, δει το θέμα αυτό η Ειδική Επιτροπή που δεν θυμάμαι και πώς τη λένε, αλλά να το μελετήσετε γιατί νομίζω ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε τη, το δικό μας, ε, τη δική μας δουλειά γιατί βρισκόμαστε σε μια αστεία πια κατάσταση. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί όλο αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη μελετήσει. Και βεβαίω θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι αυτά που πρώτα ακολουθούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και βεβαίω και τα κράτη-μέλη. Ωραία, κλείνουμε λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών για το θέμα αυτό. Πρέπει να πω ότι δεν θα είναι εύκολο για μένα να κάνω περίληψη. Θα κάνω ό,τι μπορώ πάντως. Θα βάλω τα δυνατά μου. Λοιπόν, Μιλούμε κυρίως για την ε, περιβαλλοντική αξιολόγηση που ε, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο. Λυπάμαι. Είχατε το χρόνο να παρέμβετε όπως και οι υπόλοιποι. Δεν μπορώ να σας ξαναδώσω το λόγο. Λυπάμαι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Ένα είναι αυτό και είναι το βασικό. Και θα ήθελα να αποστείλουμε μία επιστολή στην ιδιωτική εταιρεία που έχει υπογράψει τη σύμβαση και να ζητήσουμε την θέση της για τα θέματα αυτά που θίγονται στην αναφορά και κυρίως όταν πρόκειται για τα θέματα που απτούνται της σύμβασης του όρχους. Γιατί εδώ διακυβεύεται η αποτυχία της εφαρμογής όλων αυτών των διατάξεων που έχουν βεβαίω επίπτωση στην, στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Περί αυτού πρόκειται στην ε, Σύμβαση του όρχου και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πριν γίνει οποιοδήποτε βήμα ε, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τώρα, η δεύτερη σύμβαση που πρέπει επίσης να πληρείται πλήρως είναι η Σύμβαση της Φλωρεντίας και η Σύμβαση της Φλωρεντίας είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου project και δραστηριότητε που θα πρέπει να πληρούν απολύτω τι διατάξει τη συμβάση τη Φλωρεντίας πριν γίνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Οπότε θα στείλουμε στην εταιρεία την επιστολή αυτή και στι ελληνικέ αρχέ. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντο, το Υπουργείο Οικονομία, για να ζητήσουμε την άποψή του για το θέμα αυτό το οποίο θίγουν οι αναφέροντες. Και επίσης αυτό που θα πούμε στην επιστολή είναι ότι ο περιβαλλοντικός ε, έλεγχος θα πρέπει να ε, συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα πρέπει να γίνει σεβαστή η οδηγία και βεβαίως να εφαρμοστεί. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό και επιπλέον θα ήθελα ε, από καιρού εις καιρών να εμπλέκουμε και την Επιτροπή ΕΚΟΝ για το οικονομικό υποθέσεων, για το οικονομικό κομμάτι. Συμφωνείτε, συνάδελφοι. Και κάτι άλλο, ο κύριος Μαριάς. Ε, ξέρω τι θα, θα πείτε μάλλον. Μια προφορική ερώτηση θα μου πείτε, έτσι. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σε αυτή τη φάση γι' αυτό. Αυτό θα το κάνουμε στο επίπεδο των συντονιστών. Αυτό ας το συζητήσουμε σε επίπεδο συντονιστών. Εγώ θέλω να συμπληρώσω λίγο την ε, ε, πρότασή σας, διότι πρέπει να διερευνηθεί η έννοια της α, κρατικής ενίσχυσης, διότι με τα στοιχεία που θέσαμε των φοροαπαλλαγών και ταυτόχρονα όλων αυτών των κρατικών ενισχύσεων, πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Και η Επιτροπή νομίζω πρέπει να μας απαντήσει στα θέματα αυτά, αλλά να απαντήσουν συγκεκριμένα και οι ελληνικές αρχές στα συγκεκριμένα ζητήματα. Οπότε έτσι νομίζω ότι ολοκληρώνεται μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη συζήτηση και μετά σε επόμενο στάδιο που θα έχουμε όλες τις απαντήσεις θα μπορέσουμε να, να βάλουμε τα θέματα αυτά. Διότι η κυρία Κέλλερ πολύ σωστά έθεσε ένα θέμα. Αυτό που έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή μας. Πολλές φορές τη σύγκρουση συμφερόντων που έχει η ίδια η Κομισιόν ως μέλος της Τρόικας που επέβαλε αυτή την ιδιωτικοποίηση και ταυτόχρονα ως θεματοφύλακας των συνθήκων που πρέπει να ελέγξει αν τηρείται το κοινοτικό δίκαιο εν προκειμένου. Άρα λοιπόν με αυτή την πρόταση όπως την κάνατε, αν τη συμπληρώσουμε έτσι νομίζω ότι καλύπτουμε όλα τα κενά σε πρώτη φάση και μπορούμε να δούμε παρακάτω τι κάνουμε. Σύμφωνο και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τελειώνουμε τότε. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. καλό ταξίδι πίσω στην Ελλάδα και για, για τον ήλιο. Κοίταξε, πρέπει... Ε, we will, we will receive it. Do you receive it? Okay. Εντάξει, σας ευχαριστώ και θα προχωρούμε. Now we will move to a complete... Τώρα περνάμε σε μία εντελώς διαφορετική αναφορά 15-17 του 2012 και μία σειρά αναφορών, συναφών αναφορών που αναγράφονται στο σημείο 18. Είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Γιατί στις 6.30 ε, δεν θα έχουμε πια διαρμηνείς. Λοιπόν, καλωσορίζω τους αναφέροντες και σας δίνω πέντε λεπτά σε όλους. Είσαστε αρκετοί, άρα εσείς θα πρέπει να κάνετε την κατανομή. Θα μιλήσει ένας, δύο, τρεις. Θα αρχίσω εγώ. Πιέρο Βιλάντι. Εκπροσωπώ τον Στέφανο ε, Τζοβανίν. Την τελευταία φορά έγινε αναβολή ε, αντιμετώπισης της αναφοράς μέχρι ότου αποφανθεί το ΔΕΚ. Στο σημείο 43 αναφέρει το ΔΕΚ για αυτές τις εκχωρήσεις και τις αδειοδοτήσεις ότι θα πρέπει να εμπέσουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 της οδηγίας, κάτι το οποίο θα επαληθεύσει ο ε, Εθνικός Δικαστής. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, έκανε, έστειλε εξώδικο προς τις Ιταλικές αρχές, στην ουσία ανέστειλε την όλη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στα πλαίσια αυτής της απόφασης ε, ε, μιλά για τον βασικό κανόνα σε σχέση με το διάστημα εκχωρήσεων αυτών των παρακτήων χώρων μέσα στα πλαίσια μιας διαδικασίας ανανέωσης, συνεχούς ανανέωσης. για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Άρα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει το ζήτημα διαφορετικά σε σχέση με την Επιτροπή. Άρα, θα πρέπει να ε, προστατευθούν ε, οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει την αδειοδότηση. Γιατί όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει ότι σε περίπτωση αμφιβολίας για την εφαρμογή του άρθρου 12 θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 49 σε σχέση με την ελευθερία εγκατάστασης. Και σε αυτή την περίπτωση οι ε, εκχωρητές θα πρέπει να μπορέσουν να αποσβέσουν αυτή την ε, επένδυση. Και όπως μας λέει η απόφαση, θα πρέπει να εφαρμοστεί το ενωσιακό δίκαιο, ενώ οι εκχωρήσεις για τις ε, οποίες μιλάμε έχουν ε, προηγηθεί της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Επιτροπή Παόλο Λαβάντζη. Το λόγο έχει η Επιτροπή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, ο δεύτερος αναφέρω. Νόμιζα ότι είχατε τελειώσει. Καλησπέρα σας. Εμείς ε, ε, ε χωρούντες δυνάμει της οδηγίας Μπόλκεστάιν θεωρούμε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά μας το ιδιοκτησιακό μας καθεστώς και η διαδικασία εκχώρησης, διότι πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις και ε, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η εργασία είναι το μόνο έσοδο για τις ε, οικογένειές μας. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε μία αξιοπρεπή εργασία γιατί μην ξεχνάτε ότι για να λάβουμε αυτές τις άδειες υποθηκεύσαμε τα σπίτια μας. Πρόκειται για επενδύσεις που κάναμε μέχρι το 2009 και δυστυχώς δεν έγινε σωστή ερμηνεία αυτής της οδηγίας από το κράτος μας. Μιλάμε για 4.000 ε, χιλιόμετρα ως παράκτια έκθεση και γι' αυτό θα πρέπει να μην ε, αντικαθιστούμε τον ένα επιχειρηματία από έναν άλλο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ε, έμπρακτο αποτέλεσμα της οδηγίας Μπόλκεστάιν. Έχουμε να κάνουμε με μικροεπιχειρήσεις και έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας προωθώντας αυτές τις παράκτιες περιοχές γιατί μιλάμε για 4.000 ε, χιλιόμετρα ακτής που θα πρέπει να τύχουν προστασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίως η Επιτροπή συμβαδίζει με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τρία είναι τα σημεία. Η οδηγία ισχύει στην παρούσα περίπτωση ως προς τον ανταγωνισμό σε σχέση με τις εκχωρήσεις, εδώ θα πρέπει να πληρούνται δύο όροι, όπως είπαν και οι αναφέροντες. Ισχύει το άρθρο 12, υπάρχει δηλαδή ανεπάρκεια πόρων, τις οποίες θα πρέπει να υπαλληθεύσουν οι, οι εθνικές αρχές, και αν δεν ισχύει το άρθρο 12, ισχύουν οι συνθήκες που αναφέρουν ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει δύο διασυνοριακό συμφέρον κατά κάποιο τρόπο. Εμείς ευθυγραμμιζόμαστε με την θέση αυτή. Το μόνο θέμα που υπάρχει και που είναι η βάση της διαδικασίας ε, επί είναι ότι η εθνική νομοθεσία είναι οριζόντια ε, νομοθεσία. Η Ισχύει παντού. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνει μια εξέταση αναπερίπτωση. Άρα ε, τασόμαστε υπέρ της εξέτασης κατά περίπτωση. Τη στιγμή που αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με τους όρους ε, ενός ε, διαγωνισμού εκδήλωση και εκδήλωσης ενδιαφέροντος. και δεν θα πρέπει να έχουμε να κάνουμε με μια οριζόντια νομοθεσία, αλλά να αποφανθούν οι Ιταλικές αρχές αναπερίπτωση. Ε, δεν έχουμε τώρα μια Ιταλική, έχουμε μια Ιταλική υπόθεση, αλλά όχι Ιταλική επιτροπή, όπως είχαμε ελληνική πριν. Θέλει κάποιος το λόγο, έχετε το λόγο. Ε, σκουζάτε. Ζητώ συγγνώμη. Είστε ένας από τους ετούντες. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Πολύ σύντομα. Ονομάζομαι Μπέτι Φλάβιο και νομίζω ότι ερμηνεύω σωστά τα αισθήματα πολλών συναδέλφων. Εγώ έχω ένα ε, μπαρ και μικρό εστιατόριο στο Ρίμινι και έλαβα αυτή, μάλλον αγόρασα αυτό το χώρο από τον κύριο Μπέσιτς Μουσταφά σερβικής ε, καταγωγής και από όσο γνώριζα δεν υπήρχαν όρια στην είσοδο σε αυτή την αγορά των παρακτήων ε, χώρων. Όμως ε, οι Ιταλικές αρχές δεν μας επιτρέπουν που να ασκήσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και εδώ μιλάμε για μικροεπιχειρήσεις που έχουν οικογενειακό χαρακτήρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει και που την χάνουν αυτής της ε, μεταχείρισης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις ε, δημόσιες αρχές γίνονται ε, αδειοδοτήσεις οι οποίες δεν ακολουθούν διαδικασίες διαφάνειας, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η μαφία ανακυκλώνει χρήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις και μην ξεχνάμε ότι πολλοί ε, διοικητικοί υπάλληλοι έχουν συλληφθεί για παράνομες αδειοδοτήσεις στη χώρα μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι εμεί αναλαμβάνουμε τις ναυαγοσωστικές δραστηριότητες και καθαρίζουμε τις ακτές. Υπερασπιζόμαστε λοιπόν το δικαίωμα του να μπορέσουμε να σώσουμε τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Επίσης έχουμε ε, υπηρεσίες ε, πρώτης βοήθειας, πρώτων βοηθειών και προσπαθούμε να περιφρουρήσουμε τις ακτές από περιβαλλοντικές καταστροφές. Δυστυχώς όμως δεν εφαρμόζεται η οδηγία Μπόλκεστάιν. Θέλουμε να προωθήσουμε τις ακτές μας που είναι πανέμορφες. Ε, με συγχωρείτε κύριε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αποτελέσματα πριν από το τέλος της ημέρας. Στην Ισπανία εδώ και 75 χρόνια υπάρχει αυτή η διαδικασία αδειοδότησης ακολουθώντας τις αρχές της ε, ιδιοκτησίας και μπορούμε να πούμε ότι η δυνάμη του άρθρου 17 της ε, Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορούν να δράσουν. Θέλουμε να δράσει η Επιτροπή έτσι ώστε η οι κρυσταλλικές αρχές να, να συμμορφωθούν στα άρθρα 7, 16 και 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει, έχω, θα είχα πολλά να πω, αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Στην ουσία καταστρέφεται ένας οικονομικός ιστός, ο οποίος χτίστηκε εδώ και 50 χρόνια, δηλαδή μετά τον πόλεμο. Για να δημιουργηθεί μία επιχείρηση χρειάζονται πολλά χρόνια. Το να καταστραφεί ε, γίνεται σε μία στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην ουσία χαλάει, καταστρέφεται αυτός ο οικονομικός ιστός. Ελπίζω να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις επιχειρήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχουν συνάδελφοι. Έχω ένα συνάδελφο που είναι παρόν. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Εντάχει. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή, γιατί αν κατάλαβα καλά θα δεχτεί να μην ε, ληφθεί υπόψη η οριζόντια νομοθεσία, για αυτές τις παράκτιες εκχωρήσεις, αλλά να αντιμετωπίσει το ζήτημα αναπερίπτωση, όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και να μιλήσουμε βεβαίως και για τα διασυνοριακά συμφέροντα που ισχύουν από το 1984 και μετά. Ε, έχουμε εκπροσώπους από τη μόνιμη ε, αντιπροσωπεία της Ιταλίας. Ο Νίκολα Μινάτσι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους ε, συμπολίτες μας που είναι παρόντες. Εξανόματος της Ιταλικής Κυβέρνησης, το μόνο στοιχείο που θα θέλαμε να αναφέρουμε σχετίζεται με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε δύο υποθέσεις, γιατί πλέον η Ιταλία θα πρέπει να βρει έναν τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Χρειάζεται νέος νόμος και γι' αυτό είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε. Εφαρμόζοντας την απόφαση θέλουμε να υπάρξει μία εξισορρόπηση με φάση το κριτήριο του διασυνοριακού συμφέροντος και του, των ελλείψεων που υπάρχουν. Αυτή, αυτή η δραστηριότητα απασχολεί πολλές μικροεπιχειρήσεις και χιλιάδες οικογένειες και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις και οικολογικές επιπτώσεις. Άρα θα πρέπει να έχουν προστασία σε αυτές οι παράκτιες περιοχές, όπως ορίζει και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δυνάμει της εφαρμογής της οδηγίας. Από Ιταλικής πλευράς θα θέλαμε να πούμε ότι αυτή η απόφαση έχει επιπτώσεις και εκτός Ιταλίας. Μιλάμε για παράκτιες εκχωρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εφόσον λοιπόν ε, μιλάμε για τον ε, υγιή ανταγωνισμό και για το άνοιγμα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει αυτή η απόφαση να ισχύσει και να εφαρμοστεί και αλλού. Δεν θα θέλαμε η Ιταλική αγορά να ανοίξει περισσότερο από την αγορά άλλων χωρών. Χαιρόμαστε για τον ε, διάλογο με τα θεσμικά όργανα και χαιρόμαστε διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέδωσε μεγάλη σημασία στο όλο ζήτημα. Ελπίζουμε να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα και σε μία εξισορρόπηση ε, της κατάστασης σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. θα πρέπει να φτάσουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Εφόσον έχουμε μία απόφαση του δικαστηρίου, μία νοπή απόφαση, ε, δεν μιλάμε σε μία απόφαση μόνο υπέρ των αναφερόντων. Θα πρέπει να αποτιμήσουμε την κατάσταση με βάση την πρόσφατη απόφαση. Γι' αυτό θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και θα στραφούμε προς την Κομισιόν, η οποία θα αποτιμήσει την κατάσταση δυνάμει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν λοιπόν γίνει αυτή η εκτίμηση, η αξιολόγηση, θα έχουμε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα προχωρήσει. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η κυρία Μπιτζότο πρόσφατα είχε γύρει τρία ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο και δεν είχε λάβει απάντηση ακόμα. Θα πρέπει να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν στην κυρία Μπιτζότο. Όταν γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυνάμει της απόφασης του δικαστηρίου, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αυτά μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Σας ευχαριστώ όλους που ταξιδέψατε μέχρι εδώ, μέχρι τις Βρυξέλλες από την πανέμορφη Ιταλία. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή και ελπίζω την επόμενη φορά να έχει επιληθεί το θέμα των παράκτιων αυτών περιοχών. Γιατί η Ιταλία είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη, ιδιαίτερα για μας τους βόρειους και υπερβόρειους. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ και στους συναδέλφους.